Καλημέρα συνάδελφοι. Το πρώτο σημείο της ημερήσιας διάταξης αφορά τη δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις ευρωεκλογέ το 2014. Θα ήθελα να επενθυμίσω στους βουλευτές ότι για αυτή τη συζήτηση δεν προβλέπεται η διαδικασία του Eye. Δίνω το λόγο αμέσως στον Επίτροπο Σεμέτα. Έχετε το λόγο κύριε Επίτροπε. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε αξιότιμα μέλη, οι εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι πάντα πολύ σημαντικές στιγμές για την Ένωση και οι εκλογές του 2014 έρχονται σε ιδιαίτερα κρίσιμη εποχή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πάντα υποστήριζε κάθε προσπάθεια για την ενισχύση της νοημότητας του Κοινοβουλίου, όχι μόνο προς όφελος όλων των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά πάνω απ' όλα προς όφελος των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης η άμεση εκπροσώπηση είναι σημαντικό στοιχείο ε, νομιμότητας για τις δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό που χρειαζόμαστε σήμερα περισσότερο παραποτέ είναι πανευρωπαϊκές συζητήσεις, καλύτερη κατανόηση των όσων διακυβεύονται, μεγαλύτερη συμμετοχή των ψηφοφόρων και πιο άμεση σχέση μεταξύ των εκλογικών αποτελεσμάτων και της ηγεσίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στην ομιλία του το Σεπτέμβριο για την κατάσταση της Ένωσης, ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κάλεσε τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα να παρουσιάσουν τους υποψηφίους τους για την θέση του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις εκλογές του Ευρωκοινοβουλίου του 2014. Δέσμευση από τα πολιτικά κόμματα να το κάνουν αυτό το βήμα θα ενίσχυε περαιτέρω την ευρωπαϊκή διάσταση αυτών των εκλογών. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί χωρίς αλλαγή της συνθήκης, διότι η συνθήκη λέει ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο όταν προτείνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έναν υποψήφιο για πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και γι' αυτό, αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή αμέσως. Όσον αφορά την ισορροπία ανδρών και γυναικών, προωθεί ενεργά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την ισότητα των φύλων όπως ξέρετε. Όμως ζητάτε ισότητα των φύλων στο επόμενο σώμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το απευθύνεται αυτό το μήνυμα προς τον μελλοντικό πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σίγουρα θα καταλαβαίνετε ότι δεν εναπόκειται σε αυτήν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συζητήσει τι δράσει του επομένου Προέδρου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όσον αφορά τι ημερομηνίε των ευρωεκλογών το 2014, θα ήταν ατυχέ να ε, έχουμε αρνητικές συνέπειες για τη συμμετοχή στις εκλογές. Αν το Συμβούλιο προτείνει διαφορετική ημερομηνία για τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που πρέπει να τοποθετηθεί σύμφωνα με το τροποποιημένο νόμο του 1986 ε, θα πρέπει να εξασφαλιστεί η σαφήνεια, η συγκεκριμένη ημερομηνία του ταχύτερο δυνατών. Χρειάζεται ισχυρότερη πολιτική ένωση με μεγαλύτερη λογοδοσία και δημοκρατική νομιμότητα στον αφορά τι αποφάσει που λαμβάνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι και θα πρέπει να παραμείνει στο επίκεντρο όλων των συζητήσεων όσον αφορά το μέλλον τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω. Ο ρόλο αυτού του Κοινοβουλίου είναι κρισίμου σημασία στο συγκεκριμένο πλαίσιο. Σα ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ Επίτροπε. Δίνω το λόγο στους αγοριστέ εν ονόματι των ε, ομάδων των. Από το ΕΛ ξεκινάμε. Καζίνη για 1,5 λεπτό. Ο κύριος Καζίνη έχει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η πρόταση ψηφίσματος που θα ψηφίσουμε εμπεριέχει όπως είπε ήδη ο Επίτροπος τρία σημεία. Το πρώτο αφορά την πρόταξη της ημερομηνία των εκλογών. Έχει πρόθεση η πρόταση να εγγυηθεί ότι στο τέλος του καλοκαιριού ήδη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι σε θέση να ξεκινήσει τις εργασίες της θα αξιολογηθεί καλώς αν αυτό είναι εφικτό. Όπως είπε σωστά ο Επίτροπος, η ημερομηνία συνεπάγεται αύξηση της συμμετοχής. Θέλουμε να αυξήσει τη συμμετοχή σε εκλογές και μείωση. Η σημαντικότερη πρόταση όμως είναι αυτή που προβλέπει την αναφορά πλευράς πολιτικών κομμάτων. Προτιμούσα να μιλήσω για πολιτικά κόμματα παρά για πολιτικές οικογένειες για να φανεί η ανάγκη των πραγματικών σχηματισμών των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να δώσουν ένδειξη, έλεγα, για ενδεχόμενο υποψήφιο για πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτό είναι σημαντικότατο ούτω ώστε οι πολίτε, οι Ευρωπαίοι πολίτε, οι εκλογεί να ταυτιστούν με την Ευρώπη. Η μείωση τη συμμετοχή στην ψηφοφορία οφείλεται πολύ και στο γεγονό ότι κατά διάρκεια των ευρωεκλογών ε, μιλούν για άλλα πράγματα, όχι για την Ευρώπη, αλλά για εθνικά προβλήματα. Οι ευρωεκλογέ θεωρούνται ω μια επαλήθευση, αν θέλετε, των διαφόρων εσωτερικών πολιτικών ε, συζητήσεων θα πρέπει να μιλούμε για τι εκλογέ στην Ευρώπη. Θα πρέπει να πιστεύουν οι πολίτε, σοβαρά να πιστεύουν, ότι η ψήφο του μετρά όσον αφορά τι ευρωπαϊκέ πολιτικέ. Λοιπόν, πιστεύω ότι η ένδειξη του Προέδρου για τον Πρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ένα στοιχείο που δίνει αυτό το συνέστημα στου πολίτε. Θα συζητηθεί σίγουρα ε, περισσότερο το θέμα από το παρελθόν. Θα συζητηθεί περισσότερο η Ευρώπη από το παρελθόν. Διότι η οικονομική κρίση έχει ρίξει φω. Κατά πόσο χρησιμοποιούμαστε περισσότεροι ή λιγότερη Ευρώπη ή το τέλος Ευρώπης. Αυτό θα συζητηθεί. Το να δώσουμε στους πολίτες τη δυνατότητα να αποφασίσουν οι ίδιοι όσον αφορά τη διακυβέρνηση της Ευρώπης, τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι κάτι ε, απόλυτα σημαντικό. Το τρίτο θέμα αφορά τη σύνθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πέρα από το θέμα ε, των φίλων, της των φίλων. κατά πόσο θα ήταν σκόπιμο οι μελλοντικοί επίτροποι να επιλέγονται μέσω ποσοστώσεως που θα μπορούσε να καθοριστεί σαν αριθμός ή θα μπορούσε να αφαιθεί και σε κάποια αόριστη ένδειξη ε, από, μεταξύ των ερετών βουλευτών. Έτσι οι εκλογείς ε, θα μπορούσαν να αισθάνονται ότι κάτι πως μετράει η ψήφο τους. Λοιπόν, αξίζει για αυτούς τους λόγους να υποστηριχθεί το ψήφισμα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Γκουαλτιέρη για τρία λεπτά. Ο κύριος Γκουαλτιέρη έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η παρούσα κρίση δεν είναι μόνο οικονομική κρίση, είναι και μια πολιτική κρίση που συνδέεται με την αντίφαση μεταξύ της επικράτησης εθνικών πολιτικών χώρων και της απέτησης από την άλλη η Ευρώπη να έχει ευρωπαϊκή κυβέρνηση που βασίζεται επί ευρωπαϊκών θεσμών που νομιμοποιούνται δημοκρατικά σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Γι' αυτό το ψήφισμα που θα ψηφίσουμε έχει μεγάλη σημασία. Συγγνώμη. Έχω, έχω κάπως λαχανιάσει, συγγνώμη. Θα προτιμούσα να μιλήσω μετά τον επόμενο μιλητή. Δίνουμε το λόγο ε, στον κύριο Νταφ για την Άλντε που έχει το λόγο για τρία λεπτά. Uh, το πολιτικό κόμμα είναι ακριβώς ο σύνδεσμος που λείπει για την ε, διεθνική δημοκρατία. Πρέπει να αποφύγουμε την τάση που υπάρχει στη συμμετοχή και πρέπει τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα να φροντίσουμε να γίνουν εκείνα που οργανώνουν τις ε, εκλογές. Να είναι εκείνα που θα διαρθρώνουν την ιδεολογία και θα βοηθούν το κόσμο να κάνει τις πολιτικές του επιλογές ε, κατά την στιγμή της ψηφοφορίας. Η διαδικασία αυτή μπορεί να ξεκινήσει ζητώντας από τις πολιτικές μας οικογένειες να αναλάβουν την ευθύνη να χτίσουν τα θεμέλια για μια πιο ομοσπονδιακή Ευρώπη. Ο ορισμός κάποιον από τα κόμματα των πρωταθλητών τους κατά κάποιο τρόπο ως υποψήφιοι για την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όπως ε, επίσης να είναι από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οι υποψήφιοι επίτροποι είναι κάτι το οποίο ακολουθεί τη λογική της συνθήκης της Λισαβόνας. Σύμφωνα με αυτήν, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα εκλέξει και το διάδοχο του κύριου Παρόσο. Η επιτυχία μας θα κρυθεί από το πόσο θα προσωποποιηθεί και θα δραματοποιηθεί τελικά η προεκλογική εκστρατεία και κατά πόσο θα μπορέσει ο κόσμος να βάλει τη φαντασία του να δουλέψει. Τίθονται πολλά ζητήματα για το επόμενο κοινοβούλιο. Για παράδειγμα, το θέμα της ισορροπίας μεταξύ των δύο φύλων στην ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το πόσο πολύ θα εμβαθύνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στη μορφή που θα έχει ο ευρωπαϊκός προπολογισμό και βέβαια ποιο θα είναι το μέγεθος τελικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί έτσι αλλάζει η ευρωπαϊκή δημοκρατία ανάλογα με τον αριθμό των μελών και αυτό θα πρέπει να το αντιληφθούμε πλήρως και να το αντιμετωπίσουμε με εμπιστοσύνη και δύναμη. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Για τους πρασίνους, Χάφνερ για μισή λεπτά. Ο κύριος Χάφνερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η Ευρώπη δεν είναι ένα οποιοδήποτε οικοδόμημα, είναι μια δημοκρατία. Είναι η κατά τη γνώμη μας ε, και ε, η προσδοκία μας είναι να είναι μία από τις πιο σημαντικές δημοκρατίες στον κόσμο. Χρειάζεται λοιπόν ισχυρούς θεσμούς, ισχυρές αποφάσεις, αλλά εξαρτάται πώς αυτό θα μπορέσει να συνδυαστεί με τη θέληση των πολιτών. Όσο στενότερη είναι η σχέση αυτή, τόσο πιο ισχυρή θα είναι η δημοκρατία. Σήμερα πρέπει να μπορέσουμε να ενισχύσουμε τις ευρωεκλογές για να είναι ένα βασικότερο εργαλείο για εφαρμογή της ευρωπαϊκής πολιτικής. Να υπάρχει μία στενή σχέση ε, μεταξύ της επιλογής των πολιτών και της πολιτικής η οποία στη συνέχεια θα εφαρμοστεί. Οπότε ε, θα μου πείτε ε, όπως μου ελέγχθη από πού έρχεται αυτός ο κύριος Μπαρόζο πριν ε, ε, από τις ευρωεκλογές δεν είχε εμφανιστεί σαν υποψήφιος για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Βεβαίως θα μου πείτε ε, εντάξει ψηφίσατε σε ευρωεκλογές τελειώσατε. Όχι έτσι διότι στη συνέχεια υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν επηρεάζουμε και πρέπει να ενισχυθεί αυτή η σχέση και συγχρόνως θα πρέπει να υποχρεωθούν οι ευρωπαϊκές οικογένειες να γίνουν οι ευρωεκλογές όντως ευρωπαϊκές εκλογές και να μην ε, τις εκμεταλλεύονται για εθνικά θέματα. Θα πρέπει στο μέλλον οι πολιτικές οικογένειες πρώτων εκλογών να μας έχουν πει ποιος είναι ο υποψήφιός τους για την θέση του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του πιο ισχυρού οργανισμού μέσα στο ευρωπαϊκό αυτό οικοδόμημα να υπάρξουν πολιτικές πλατφόρμες να μπορέσουν να παρουσιαστούν τα οράματά τους για την Ευρώπη στο μέλλον ε, κατά τρόπον ώστε να ενισχύσουμε την νομιμοποίηση αλλά και την αντιπαράθεση πολιτικά μεταξύ των θέσεων που διέπουν την Ευρώπη κατά τρόπον ώστε ο πρόεδρος ή η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατόπιν αυτών των εκλογών να ε, επιλεγούν από από την αριστεία που προέκυψε από τις εκλογές. Στο μέλλον θα θέλουμε τουλάχιστον το ίμιση ε, τουλάχιστον των επιτρόπων να προέρχεται από το Ευρωκοινοβούλιο κατά τρόπον ώστε να ανταποκρίνονται στη θέση ε, των πολιτών και να ενισχύσουν την ευρωπαϊκή πολιτική. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για το ECR. Κύριος Φόξ για 1,5 λεπτό έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον κύριο Κασίνη και τα, τους συναδέλφους μέλη της Επιτροπής για τη δουλειά που έκανε για το ψήφισμα. Περιέχει αρκετές καλές συστάσεις. Συμφωνούμε όλοι ότι πρέπει να βελτιώσουμε τις διαδικασίες των επομένων ευρωπαϊκών εκλογών. Θα πρέπει να ενθαρρύνουμε μεγαλύτερη συμμετοχή στις εκλογές από πλευράς πολιτών μας. Υποστηρίζω την προτινόμενη αλλαγή, δηλαδή να προταχθούν οι εκλογέ από Ιούνιο στο Μάιο 2014. Αυτό θα επιτρέψει το Κοινοβούλιο περισσότερο χρόνο για να ελέγξει τον νέο Πρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και στον Ηνωμένο Βασίλειο η διεξαγωγή των εκλογών τον Μάιο θα διευκολύνει τη διασύνδεση των ευρωπαϊκών εκλογών με τι δημοτικέ εκλογέ και αυτό θα εξοικονομήσει χρήματα του προλογωμένου και θα αυξήσει, φαντάζομαι, τη συμμετοχή. Ε, χαίρομαι για αυτήν την παράγραφο που ζητά τουλάχιστον οι μισή επίτροποι να προέρχονται από μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που αφαιρέθηκε από την Επιτροπή. Δεν θα πρέπει να ε, περιορίσουμε το δυνατότητα των κρατών μελών να επιλέξουν ποιοι θέλουν να είναι επίτροπο. Ελπίζω η Νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή να και άνδρε και γυναίκε με πραγματικά ταλέντα. Θα πρέπει να διορίζονται βάσει των προσόντων του και μόνο, τη αξία του. Δεν υποστηρίζω το αίτημα που έχει έκθεση ότι τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα να καθορίζουν υποψήφιο για τον θέση του Προέδρου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή που θα πρέπει να ηγηθεί τη εκστρατεία. Τα κράτη-μέλη στο Συμβούλιο επιλέγουν τον νέο Πρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ρωτώ το εξή ερώτημα πλευρά για του συναδέλφου. Αν τα και το δεξιά κόμματα έχουν πλειοψηφία στο Συμβούλιο 2014, πραγματικά πιστεύετε ότι θα διορίσουν σοσιαλιστή ίσως σαν τον Μάρτιν Σούλτς να είναι πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μόνο διότι τα σοσιαλιστικά κόμματα έχουν περισσότερες ψήφους από το ΕΛΚ σε ευρωεκλογέ. Κατά την άποψή μου αυτό δεν θα συμβεί και γι' αυτό το λόγο η ομάδα μου δεν μπορεί να υποστηρίξει αυτό το ψήφισμα. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ ε, ε, για την ομάδα του ο κύριο Άγνιου. Όχι. Δεν είναι δυνατόν ούτε γαλάζια κάρτα, ούτε catch the eye. Εξετάσαμε τον κανονισμό από αυτού. Λοιπόν, ε, ο κύριος Άκνιου για ένα λεπτό έχει το λόγο. Ε, ε, λοιπόν, δίνω το λόγο στο κύριο Γκουαλτιέρη, όχι μετά. Καλώς. Το επόμενο όνομα που έχω μπροστά μου είναι Σόνενγκάρτ για την ΚΟΥΕ για δύο λεπτά. Κύριο Σόνενγκάρτ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η ομάδα μας υποστηρίζει την διεκδίκηση αυτή για την κατανομή μεταξύ ανδρών και γυναικών ε, στην Επιτροπή ακόμα και αν αυτό δεν το πετύχουμε στην επόμενη Επιτροπή, είναι κάτι που πρέπει να το πάρουμε πολύ στα σοβαρά και να αντικατοπτρίζεται στα όργανά μας. Αλλά ό,τι θετικό και αν έχω να πω για το ψήφισμα αυτό τελειώνει εδώ. Γιατί μετά έχουμε την πρόταση για τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα που θα πρέπει, λέει, να ορίσουν τον υποψήφιο για την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Με το ερώτημα τίθεται από πού ξεκινάει αυτή η ιδέα είναι κάτι το οποίο έχουν εκφράσει λέει της Ευρώπης, είναι κάτι το οποίο έχουμε διαβάσει σε κανένα σύνθημα στις διαδηλώσεις που έγιναν στην Αθήνα, τη Μαδρίτη, τη Λισαβόνα. Όχι. Έρχεται από πάνω η πρόταση αυτή, από τον Παρόσο ο οποίος ε, το είπε στην ομιλία του που έκανε για την κατάσταση τη Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ στο Κοινοβούλιο. Αλλά η δημοκρατία πρέπει να ξεκινάει από κάτω, από τη βάση. Και αν τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα θέλουν να παρουσιάζουν υποψηφίου για την Προεδρία τη Ευρωπαϊκή Επιτροπής, α το κάνουν. Εντάξει, φυσικά και γίνεται. Υπάρχει δυνατότητα αυτή. Ό,τι γνώμη και να έχουμε για τον Παρόσο ε, και ό,τι και λέει και ο Παρόσο. Υπάρχει έλλειμμα δημοκρατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν θα το ε, λύσουμε αν ε, προσωποποιήσουμε την ε, συζήτηση αυτή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Χρειαζόμαστε περισσότερη δημοκρατία και γι' αυτό η ομάδα μας έχει υποβάλει πρόταση που καλεί τα κράτη-μέλη να παρουσιάσουν ένα εκλογικό σύστημα το οποίο να διασφαλίζει ότι τα πολιτικά κόμματα με αναλογικότητα εκπροσωπούνται στις εκλογές αυτές. Γιατί τι να την κάνουμε μια δημοκρατία η οποία αποκλείει κάποια κόμματα, την άποψη δηλαδή κάποιων ανθρώπων. No taxation without representations, όπως έχουμε ακούσει τόσες φορές. Αυτή λοιπόν ε, η πρόταση δεν δικατοπτρίζει τις δημοκρατικές ε, απαιτήσεις και είναι κάπως περίεργο γιατί όπως ε, είπα η Ευρώπη δεν χρειάζεται περισσότερη προεδρία, χρειάζεται περισσότερη δημοκρατία. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ο λόγος στον κύριο Γκουαλτιέρη για τρία λεπτά. Ευχαριστώ, ευχαριστώ Πρόεδρε. Έλεγα, λοιπόν, ότι η κρίση που περνά το ευρώ δεν είναι απλώς οικονομική κρίση, αλλά είναι πολιτική κρίση επίση που απορρέει από μια αντίφαση όλο και πιο μεγάλη μεταξύ της επικράτησης εθνικής διάστασης που ισχύει ακόμα της πολιτικής και του ευρωπαϊκού χαρακτήρα των απαραίτητων πολιτικών για την αντιμετώπιση της κρίσης από την άλλη. Λοιπόν, η μεταρρύθμιση που αυτό το ψήφισμα προτείνει να ελοπιθεί μια μεταρρύθμιση που δεν απαιτεί τροποποίηση των συνθήκων, δεν απαιτεί τροποποίηση της δευτεροβάθμιας νομοθεσίας, αλλά είναι μεγάλη όμως πολιτική και θεσμική μεταρρύθμιση, διότι μέσω του σύμφωνα με το κοινοβουλευτικό καθεστώ. Δεν μιλάμε για άμεσε εκλογέ, μιλάμε για το μοντέλο των κοινοβουλευτικών δημοκρατιών. Μέσω του μηχανισμού τη πρόταση από πλευρά πολιτικών κομμάτων, ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων, που είναι αναγνωρισμένα από τι συνθήκε, είναι μια οντότη που εκπροσωπεί τι συνθήκε, να προτείνουν κάποιον υποψήφιο για την Προεδρία τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όχι μόνο εφαρμόζει το πνεύμα και το γράμμα των συνθήκων που λένε ότι η Πρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκλέγεται από το Κοινοβούλιο και ότι ο καθορισμός του θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη το αποτέλεσμα των εκλογών αλλά υλοποιεί και μία μεταρρύθμιση η οποία επιτρέποντας στους πολίτες να συμμετέχουν άμεσα στην επιλογή της πολιτικής κυβέρνησης Ευρώπης προσφέρει αυτή την ομιμοποίηση τη δημοκρατική που εδράζεται επί αυθεντικού ευρωπαϊκού πολιτικού χώρου στους κοινούς θεσμούς που ε, ε, επηρεάζει την κυβέρνηση τις πολιτικές δράσεις και πέρα από τη δημοκρατική νομιμοποίηση που δίνει στις πολιτικές. Απ' την άλλη αυτή η μεταρρύθμιση κατά την άποψή μου δεν είναι καθόλου ε, σε σύγκρουση με τον ανεξάρτητο χαρακτήρα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διότι το άρθρο 17 το οποίο αναφέρεται στην ανεξαρτησία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το βαθμό στον οποίο αναφέρεται σε ειδική πλειοψηφία στο Συμβούλιο και αναφέρεται στα αποτελέσματα των εκλογών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δείχνει αυτό το άρθρο σαφώς όπως γίνεται και στα συνηθισμένα δημοκρατικά καθεστώτα ότι η νομιμοποίηση, η δημοκρατική και η ανεξαρτησία ενός οργάνου κυβερνητικού ε, δεν βρίσκονται αυτά τα δύο που ανέφερα σε αντίφαση. Εκδημοκρατικοποιείται η δράση, ενισχύεται η δράση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και συνεπώς δημιουργείται μια Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι πιο νόμιμη, πιο ισχυρή, πιο κοντά στους πολίτες και πιο ικανή να δώσει απαντήσεις στην, στην φοβερή αυτή κρίση που αντιμετωπίζουμε και που με τέτοιε μεταρρυθμίσεις μπορεί αυτή η κρίση να γίνει και μια δυνατότητα για να κάνουμε άλλο ένα βήμα προόδου όσον αφορά το δρόμο για την Ευρωπαϊκή για την πολιτική Ευρώπη. Ευχαριστώ κύριε Σιγκλέρ, διαδικαστικό. Ορίστε. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Είναι πολύ ηρωνικό όταν συζητάμε περί δημοκρατίας ότι ε, αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταστέλει τη συζήτηση χωρίς ε, την χρήση μπλε κάρτας ή catch the eye και όλοι βεβαίως θα είμαστε υποψήφοι για το 2014 σε ευρωεκλογές. Μας είπατε ότι ε, δεν θα υπάρχει catch the αλλά ποτέ δεν είπατε προηγουμένως ούτε στη γραπτή μας επικοινωνία ότι δεν θα υπάρχει μπλε κάρτα και βλέπετε ότι η Ευρώπη μιλάει για δημοκρατία χωρίς όμως να την εφαρμόζει πρακτικά. Σας ευχαριστώ κυρία Σινκλέρ. Εγώ είπα στην αρχή ότι δεν προβλεπόταν η διαδικασία προσέγγισης προσοχής του Προέδρου διότι αυτή ήταν ε, η συμφωνία των πολιτικών ομάδων τη Δευτέρα, διότι το σημείο ενετάχθη στην ημερήσια διάταξη τη Δευτέρα. Στην πράξη ουσιαστικά μιλά μόνο για ένα βουλευτή πάρει το λόγο της ομάδας του. Η ομάδα των μη εγγεγραμμένων δεν ζήτησε να παρέμβει και όμως είναι στη διοικητική ευχαίρεια του Προέδρου να δώσει τη δυνατότητα παρέμβασης με τη γαλάζια κάρτα. Δίνω το λόγο τώρα στον Επίτροπο Σεμέτα. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, αξιότιμοι ευρωβουλευτές. Όπως είπε και ο πρόεδρος Βαρόσο όταν απευθύνθηκε στο Κοινοβούλιο επί τη ευκαιρία της συζήτησης για την κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χρειαζόμαστε έναν ευρωπαϊκό χώρο που να συζητούνται και να προβληματιζόμαστε πάνω στα ευρωπαϊκά θέματα. Δεν μπορούμε να περιμένουμε ότι θα λύσουμε τα ευρωπαϊκά προβλήματα σε εθνικές συζητήσεις και προβληματισμούς. Και νομίζω ότι είναι σωστό αυτό. Γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιστεύει ότι η δικιά σας συμβολή για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής πολιτικής διαδικασίας είναι κάτι θετικό γιατί έτσι και οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορούν να δραστηριοποιηθούν περισσότερο και να συμμετέχουν ενεργά. Στις εκλογές, για παράδειγμα, του 2014, αλλά και μετά από αυτές. Η ιστορία με τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα που θα μπορούν να υποβάλουν ε, τις υποψηφιότητες για την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πιστεύουμε ότι θα αποτελέσει ένα σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Για την επιλογή των επιτροπών, το πιο σημαντικό είναι οι επίτροποι αυτοί, οι υποψήφοι, να επιλέγονται βάσει των ικανοτήτων τους, βάσει της δέσμευσής τους υπέρ της Ευρώπης και βάσει της ανεξαρτησία τους. Εξάλλου η συνθήκη προβλέπει ένα συγκεκριμένο μηχανισμό για την επιλογή των επιτρόπων. Στα πλαίσια αυτά λοιπόν, οι ευρωπαϊκές πολιτικές οικογένειες είναι πάντα ελεύθερες να ψάξουν να βρουν τον καλύτερο τρόπο για να διασφαλίσουν τους καλύτερους υποψηφίους. Όπω και να έχει το πράγμα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ακροάσει, οπότε έρχονται οι επίτροποι, ε, συζητάει το Κοινοβούλιο μαζί του και αποφασίζει. Και υπάρχουν και άλλα στοιχεία όπου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα αλλά και χώρε μέλη μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να προωθήσουν την ευρωπαϊκή ιδέα και να την κάνουν ακόμα πιο ελκυστική για του πολίτε μα. Τώρα είναι κατάλληλη στιγμή για να πάρουμε τις αποφάσεις που πρέπει θαραλές εν ώψη των ευρωεκλογών του 2014. Με αυτό το πνεύμα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υποβάλει τις προτάσεις της για να ενισχύσει την δημοκρατική νομιμότητα της Ευρωπαϊκής μας Ένωσης. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ Επίτροπε. Λάβαμε μια πρόταση ψηφίσματος. Η συζήτηση περατώθηκε, η ψηφοφορία θα λάβει χώρα σήμερα στις 12. Τώρα στην ημερήσια διάταξη έχουμε την παρουσίαση της ετήσιας εκθέσεως. Έλεγα λοιπόν ότι προβλέπεται η παρουσίαση της ετήσιας εκθέσεως για το 2011 του ελεγκτικού συνεδρίου αλλά περιμένουμε τον πρόεδρο Οπότε περιμένουμε κάποια λεπτά.